ή Οι τίτλοι θα δημοσιευθούν στα πρακτικά αυτής τη συνεδρίασης. Περνάμε τώρα στο πρόγραμμα εργασία αυτής της εβδομάδα. Έχουμε το, το σχέδιο μερίσιας διάταξη το οποίο εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 137. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση αλλαγής για σήμερα. Περνάω στην τρίτη. ομάδα του ΕΛΚ ζητάει προφορικό ερώτημα προς την Κομισιόν για τη διακριτική μεταχείριση των τελωνίων ε, στα ρωσικά σύνορα των τελωνίων με πινακίδες Λιθουανίας. Ποιος θα ήθελε το λόγο εδώ πέρα, ο κύριος Κάσπαρη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εδώ και λίγες ημέρες έχουμε την εξής ε, κατάσταση. Οι ρωσικές αρχές σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω αυθαιρετούν εις βάρος ε, φορτηγών από την ε, Λιθουανία τους αναγκάζουν τους οδηγούς να ξεφορτώσουν όλο το φορτίο και να το ξαναφορτώσουν. Είναι καψόνια εν ώψη της ε, συνόδου κορυφής, της προσεχούς συνόδου κορυφής. Και χωρίς να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από σήμερα το μεσημέρι απαγόρευσαν την εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από την Λιθουανία. Είναι απαράδεκτο η Ρωσία να ε, συμπεριφέρεται έτσι με αυθαίρετα μέτρα εις βάρος της ε, χώρας ε, η οποία αυτή τη στιγμή ασκεί την Προεδρία. Και θα θέλαμε να απευθύνουμε ερώτημα προς την Κομισιόν. Το έχουμε επεξεργαστεί με πολλούς ε, συναδέλφους από την Επιτροπή Εξωτερικών Θεμάτων και θα θέλαμε τη στήριξή σας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φόβοντα θα ήθελε να στηρίξει το αίτημα αυτό. Παρακαλώ. Το στηρίζουμε πλήρως. Είναι σκανδαλώδε το πώς συμπεριφέρεται στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ρωσία. Ειδικά αν δούμε και το τι κάνει η Λιθουανία ε, και πιστεύω αυτό σχετίζεται με τη Σύνοδο Κορυφής ε, στο Βιλνίους ε, της Ανατολικής Γειτονίας. Ανάλογα πράγματα συμβαίνουν και με Ουκρανία και με Μολδαβία. Σπάνε τα νεύρα των ανθρώπων εκεί πέρα και βλέπουμε πραγματικά αυτή την συμπεριφορά τα καψόνια που γίνονται εις βάρος των οδηγών αυτών των φορτηγών. Και οπωσδήποτε είμαστε υπέρ της ερώτησης αυτής. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ε, θα ήθελε να λάβει τον λόγο εναντίον ε, του ερωτήματος αυτό. Όχι. Ωραία. Οπότε θα ψηφίσουμε το έτοιμο αυτό στην, την τρίτη το απόγευμα δηλαδή να ε, προσθεθεί το θέμα αυτό. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Οπότε εγκρίνεται και μπαίνει στη μέρη διάταξη. Για την τρίτη. Κυρία Τσίμερ, παρακαλώ. Ναι, για την τρίτη. Για την ψηφοφορία. Ρωτήσατε ποιος είναι υπέρ και μετά είπατε εγκρίνεται και να μπει μετά τις εμπορικές σχέσεις με την Ταϊβάν. Θα ήθελα όμως να πω το εξής. Έχουμε με αυτόν τον τρόπο το εξής φαινόμενο. Ο χρόνος εργασίας των πιλότων θα πάει ακόμη πιο μετά. Θέλω να το αλλάξουμε για να συζητηθεί το θέμα αυτό σε μια χρονική στιγμή στην οποία θα μπορεί και να αντιδράσει κάποιος ε, ε συνάδελφος. Έχετε δίκιο κυρία Τσίμερ. Πράγματι το θέμα που αναφέρατε πάει πιο πίσω έτσι, αλλά δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να πάει αυτό το θέμα. Ε, εκεί πέρα ζητήθηκε να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Λυπούμε. Τετάρτη, η ομάδα του ΕΛΚ προτείνει να αλλάξει ο τίτλος ε, της συζήτησης μεταναστευτικής πολιτικής ε, μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο. Και θα πρέπει να λέγεται ως εξής δήλωση του Συμβουλίου και της Κομισιόν για τις μεταναστευτικές ροές ε, στη Μεσόγειο με ε, ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα της ε, Λαμπεντούζας. Τον λόγο ζήτησε η ομάδα του ΕΛΚ, δεν ξέρω ποιος ακριβώς. Ναι, ο κύριος Γιακολίνο. Μάλιστα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, όπως υπενθυμίσετε και εσείς πριν λίγο, 200 θύματα έχουν ε, προς το παρόν μαζευτεί από τη Λαμπεντίζα και ο κατάλογος ε, δυστυχώς φαίνεται ότι θα γίνει πολύ μεγαλύτερος. Υπολογίζουμε περίπου 350 νεκρούς. Ε, ε, μία τραγωδία, ένα βήμα από το νησί. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζητήσαμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση η οποία γίνεται την ίδια ημέρα την οποία ο πρόεδρος Μπαρόζο με την Επίτροπο Μάλστρομ δικαίως θα μεταβούν στο νησί προκειμένου να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους ε, και τη βοήθειά τους και όπως αρμόζει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον αυτών των ανθρώπων ε, και της περιοχής. Ζητούμε λοιπόν να γίνει και ένα βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή η συζήτηση θα μπορούσε ίσως να γίνει στις 5, όπως ενδεικτικά είχε προβλεφθεί, για να υπάρχει παρουσία όπως ε, πρέπει του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μπαρόζο και της Επιτρόπου Μάλστρομ και του Συμβουλίου. Αύριο ε, παρουσία της Επιτροπής θα συζητηθούν αυτά τα θέματα και ελπίζουμε ότι αυτά τα οποία θα κάνουν ε, θα είναι βάσει των αρχών της αλληλεγγύης τις οποίες επιθεμούμε συνεχώς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιακορίνο. Ποιος υποστηρίζει αυτή την πρόταση, ο κύριος Σουμπαμποντα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποστηρίξω αυτή την πρόταση γιατί είναι πολύ σημαντικό η συζήτηση να γίνει παρουσία του ε, Πρόεδρου κυρίου Μπαρόσο και της κυρίας ε, Μάλστρομ. Όλη η Ευρώπη θα πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς που χάνουν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Αλλά Πρέπει να σταματήσει και η προσπάθεια κολασμού των ψαράδων που τους έχουν βοηθήσει για να σώσουν τη ζωή τους. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν αυτή η νομοθεσία στην Ιταλία. Όσοι βοηθούν τους ανθρώπους αυτούς που κινδυνεύει η ζωή τους, δεν είναι δυνατόν όπως έχει η νομοθεσία σήμερα στην Ιταλία να τιμωρούνται και να αντιμετωπίσουν ποινικέ ευθύνε. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσω και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με τον κύριο Μπαρόσο και την κυρία Μάλστρομ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κάποιος εναντίον της πρότασης θα ήθελα να λάβει το λόγο. Κυρία Χάμς, είσαστε εναντίον. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Χάμς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Από ό,τι ξέρω, το έχουμε ανακοινώσει. Η ομάδα μου φυσικά υποστηρίζει την πρόταση αλλαγή του τίτλου. Αλλά επειδή ανέφερε κάτι ο κύριος Φόμποντα από την Süddeutsche Zeitung για τα κροκοδίλια δάκρυα και να δούμε αν τελικά όλα αυτά γίνονται μονάχα σε φραστικό επίπεδο ή αν είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει. Εμεί θα θέλαμε να προσθεθεί και ένα ψήφισμα στο σημείο αυτό τη τη διάταξη. Ωραία, κυρία Χάμς. Η πρόταση είναι να γίνει αυτή η συζήτηση μαζί με ψήφισμα που θα τη συνοδεύει. Ωραία. Για την... Ε, προς το παρόν δεν έχω καμία... Μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή. Υπάρχει λοιπόν συμφωνία για την συζήτηση με το Συμβούλιο και την ε, Κομισιόν για το θέμα μετανάστευσης μαζί με, την, ε, με το δράμα της Λαμπεδούσα. Η κυρία Χάμς πρότεινε αυτή η συζήτηση να γίνει μαζί με την κατάθεση και την ψήφιση ψηφισμάτων. Ο κύριος Γιακολίνο θέλει το λόγο σχετικά. για να επιβεβαιώσω αυτά τα οποία είπε λίγο και ο συνάδελφος ε, Σβόμποντα. Είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε αυτό, αλλά δεν θα πρέπει εδώ να αμφισβητούμε την νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους. Εδώ δεν είναι θέμα νομοθεσίας κρατών μελών, είναι θέμα ε, καταμερισμού των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων. Είμαστε υπέρ τη συζήτηση, αλλά δεν θεωρούμε ότι σήμερα είναι κατάλληλη στιγμή για ένα ψήφισμα το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει εντάσει. Διότι στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν θέλουμε ούτε εντάσει, ούτε διαμάχε, αλλά πρέπει να είναι ενωμένο όλο το Κοινοβούλιο. Αυτό το ερμηνεύω σαν μια ε, θέση κατά του ψηφίσματος, κατά της συνοδείας με ψήφισμα της συζήτηση αυτής. Λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Χάμ ζήτησε να υπάρχει και ένα ψήφισμα. Ο κύριος Γιακολίνο είπε ότι δεν θέλει ένα τέτοιο ψήφισμα. Η κυρία Τσίμερ θέλει να μιλήσει υπέρ της προσάρτηση ψηφίσματος, μάλιστα. Θέλω να υποστηρίξω την πρόταση της κυρίας Χάρμς να κλείσει η συζήτηση και το σημείο αυτό τη ημερήσια διάταξη με ένα ψήφισμα, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πούμε συγκεκριμένα τι θέλουμε να αλλάξει. Αυτό ο, με το βλέπουμε στραμμένο όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσει αυτή η απάνθρωπη μεταχείριση των ατόμων αυτών που προσπαθούν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία λέει ο πρόεδρος. Θα πρέπει να ψηφίσουμε τώρα για την αλλαγή. Κύριε Σφόμποντα χωρίς μικρόφωνο. Προτείνω να γίνει αυτό το ψήφισμα στην δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Δεν μπορούμε όταν έρχεται ο πρόεδρος του, της Κομισιόν και παρουσιάσει τα θέματα αυτά να μπορούμε αμέσως εμείς να ψηφίσουμε ένα ψήφισμα. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό όμως τη ψήφιση του τελικού ψηφίσματος για τη συζήτηση αυτή στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου σε δύο εβδομάδες. Ωραία, επανέρχομαι να ψηφίσουμε καταρχήν για το αν το θέμα αυτό θα τεθεί στη μέση διάταξη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ωραία. Ομόφωνα έχει αποφασιστεί η εγγραφή του σημείου αυτού στην ημερήσια διάταξη. Τώρα έχουμε δύο διαδικαστικές προτάσεις. Ή ψήφισμα αυτή τη βδομάδα ή ψήφισμα στη δεύτερη βδομάδα ολομέλειας του Οκτωβρίου στο φως των πληροφοριών που θα μας δώσει ο κύριος Μπαρόσο και η κυρία Μάρσουμ. Κυρία Χάρμς, έχετε το λόγο. Μπορούμε να συμφωνήσουμε εάν θέλουμε να λάβουμε υπόψη όλα αυτά που θα πει ο πρόεδρος της Κομισιόν και η κυρία Μάστον, μπορούμε να κάνουμε το ψήφισμα στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Έχω λοιπόν μόνο μία πρόταση μονάχα για το ψήφισμα τη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Υπέρ, κατά, αποχές και αυτό έχει αποφασιστεί. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Για Τετάρτη δεν έχω κάποια άλλη προτινόμενη αλλαγή. Πέμπτη, οι πράσινοι ζητούν μια δήλωση τη Κομισιόν για την σύλληψη ακτιβιστών της Greenpeace στη Ρωσία σαν πρώτο σημείο την ημερήσια διάταξη της Πέμπτης και στη συνέχεια να ακολουθήσει ένας γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες. Ποιος θέλει να αιτιολογήσει αυτή την πρόταση, κύριε Χάμς. Όταν προετοιμάσαμε αυτή την αίτηση, υπήρξε ο φόβος όταν συζητούσαμε τις άλλες ομάδες ότι είχαμε πάρα πολλά σημεία τα οποία είχαν να κάνουν με τη Ρωσία και κατά την άποψή μου πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ στεναροί σε σχέση με το ρόλο της Greenpeace που είναι ένας μεγάλος μη κυβερνητικός οργανισμός σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την εργασία τους στην Ρωσία. Θυμάστε όλα αυτά που έγιναν με το Rainbow Warrior, τώρα τα ίδια έχουν γίνει με το Arctic Sunrise. Είναι απαραίτητο να ξέρουμε ότι είναι απαραίτητο να προασπίσουμε τη δυνατότητα της Greenpeace να κατεβαίνει σε δράσεις οι οποίες είναι ειρηνικές υπέρ των, της προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν μπορεί αυτό να θεωρηθεί ότι είναι μια μορφή πειρατεία σε καμία περίπτωση. Επομένως και εδώ θα πρέπει να υποστηρίξουμε την Greenpeace. Θέλω να κάνουμε λοιπόν μια συζήτηση για το θέμα αυτό την ε, Πέμπτη και να συνοδεύεται αυτή η συζήτηση από ένα ψήφισμα στη δεύτερη όμως Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο για το θέμα αυτό. Κατά. Κύριε Μακίνη, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρωτού λάβω το λόγο εναντίον. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Εμείς δεν διαφορούμε με τη σημασία αυτού του θέματος ότι αφορά την Greenpeace και τη Ρωσία. Να αναφέρω όμως στους συναδέλφους ότι την Πέμπτη το πρωί υπάρχει μια προφορική ερώτηση ήδη για το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση έχουμε κάθε ευκαιρία να γύρουμε τα θέματα που είναι σημαντικά σε σχέση και με την Greenpeace. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μακίνες. Μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα σε σχέση με την πρόταση των Πρασίνων. Ποιο υποστηρίζει Δηλαδή η πρόταση αυτή είναι να υπάρξει μια δήλωση τη Κομισιόν για του ακτιβιστέ τη Greenpeace σαν πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Ποιο υποστηρίζει την πρόταση των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Ποιο είναι κατά. Αποχέ. Από ό,τι βλέπω είναι αν θέλετε να ελέγξουμε, βέβαια, αν νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 71 υπέρ, 101 κατά. Ωραία. Κύριε Μακίνες, αν θέλετε να αιτιολογήσετε την εναλλακτική σας πρόταση τώρα. Ήθελα να με σαφείς ότι θα έπρεπε το σημείο αυτό να ενσωματωθεί στη συζήτηση για το προφορικό ερώτημα που αφορά τη Ρωσία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορεί να δεχτεί η Ολομέλεια λοιπόν την πρότασή μου ώστε να γίνει το θέμα αυτό τμήμα της συζήτηση που θα κάνουμε ούτως ή άλλως την Πέμπτη το πρωί. Äh, Κύριε Μακίνες, κατανοώ την πρόθεσή σας, αλλά την Τετάρτη αντιμετωπίζουμε άλλα πράγματα. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κυρία Χάμς, μπορούμε τότε να συμφωνήσουμε. Αν δεν θέλουμε να υπερφορτώσουμε τα ζητήματα για τη Ρωσία, να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε 14 μέρες για το θέμα αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτούς που προετοιμάζουν την ε, αγωγή στο Διεθνές Δικαστήριο σε σχέση με την περίπτωση της ΔΡΙΝΣΠΑΚ ε, και για όλους αυτούς που έχουν συμπατριώτες τους οι οποίοι είναι κρατούμενοι στο Μουρμάνσκ. Ωραία. Θα θέσουμε το σημείο αυτό στην ε, ε, στο σχέδιο ημερήσια διάταξης που θα έρθει στην ε, συνέλευση των Προέδρων και μπορούν να αποφασίσουν οι πολιτικές ομάδες για το αν θέλουν ή όχι να το εγγράψουν ημερήσια διάταξη. Εντάξει. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να το λόγο. Όχι. Έχει αποφασιστεί λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Ερχόμαστε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι μια προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν σε σχέση με την αγορά διοξιδίου του άνθρακος το 2012.